Επόμενο σημείο της ε, ημερήσιας ε, διάταξης είναι οι δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης και 26ης Ιουνίου και η συνάντηση κορυφής ε, εχθές, η συνάντηση της Eurogroup. Το λόγο θα ήθελα καταρχήν να δώσω στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον κύριο Τούσκ.